Το επόμενο θέμα στην ημερήσια διάταξη είναι η ώρα των ερωτήσεων προς το Συμβούλιο και θα ασχοληθούμε με τις ερωτήσεις που έχουν κατατεθεί για το Συμβούλιο. Η πρώτη ερώτηση σήμερα στην ε, ημερήσια διάταξή μας προέρχεται από τον κύριο Παπα-Νικολάου και αφορά τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας στο θέμα της, στον τομέα της λαθρομετανάστευσης. Έχετε το λόγο. Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, όπως γνωρίζετε, η ενίσχυση της συνεργασίας με τι τρίτες χώρες, προέλευση ή διέλευση μεταναστών, είναι βασικό στοιχείο για την μάχη της Ένωσης κατά της παράνομης μετανάστευσης. Αυτό ήταν και μία από τις μεγάλες αλλαγές και εξελίξεις που διαπιστώθηκαν μετά από αυτό που αποκαλέσαμε ως ε, σφαιρική αντιμετώπιση για τη μετανάστευση και του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη μετανάστευση και το άσυλο. Την σημασία της συνεργασίας Είναι, δεν σας ακούει, δεν ακούτε, ακούγεται ελληνική διερμηνία. Δεν ξέρω αν ακούτε. Ακούγεται η ελληνική Ακούτε την ελληνική διερμηνία τώρα. Για μίλεση. Ακούτε παρακαλώ κύριε Παπα-Νικολάου. Μας ακούτε. Είμαστε στο κανάλι. Πρέπει να βρείτε το ελληνικό κανάλι. ακούγονται τα ελληνικά παρακαλούμε. Κύριε Υπουργέ, αν μπορείτε να ξαναρχίσετε. Μήπως μπορείτε να ξαναρχίσετε την απάντησή σας για να ακούσει την ερώτηση από την αρχή ο ερωτών. Ευχαριστώ. Έλεγα κυρία Πρόεδρε ότι η συνεργασία με τρίτες χώρες είτε προέλευσης είτε διέλευσης μετανάστευσης είναι ένα από τα βασικά και πιο σημαντικά στοιχεία της νέας πολιτικής μετανάστευσης. Πριν το 2004 δεν υπήρχε στην πραγματικότητα μια ευρωπαϊκή πολιτική μετανάστευσης. Η πολιτική αυτή εμφανίζεται μετά την συνάντηση του Χάμπτον και το 2004 και ένα από τα πρώτα της στοιχεία είναι η συνεργασία με τις χώρες προέλευσης και διέλευσης παράνομης μετανάστευσης. Τούτο, όπως έλεγα, αποτελεί τμήμα του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Προς την κατεύθυνση αυτή, ήδη στα συμπεράσματα του Δεκεμβρίου πέρυσι για την διεύρυνση, το Συμβούλιο εξέφρασε την ικανοποίησή του για το ξεκίνημα του ενισχυμένου διαλόγου για τη μετανάστευση με την Τουρκία και ζήτησε την υιοθέτηση συγκεκριμένων μέτρων, για παράδειγμα την επανεισδοχή, ελέγχου στα σύνορα κτλ. Το πρόγραμμα της Στοκχόλμης επανεπιβεβαίωσε την ανάγκη αυτή δράσης κατά της λαθρομετανάστευσης. Επιπλέον δε είναι σαφές ότι το πρόγραμμα της Στοκχόλμης τονίζει όπως και το συμπεράσμα του Συμβουλίου το Δεκέμβριο του 9, τονίζουν ότι θα πρέπει να συναυθεί το συντομότερο δυνατό μια σειρά συμφωνιών ε, επανεισδοχής με την Τουρκία και η επιβεβαίωση μεταξύ εφαρμογή των υφιστάμενων συμφωνιών. Ο τελευταίο γύρο διαπραγματεύσεων, μπορώ να σα πω, έλαβε χώρα για την ε, συμφωνία αυτή επανεισδοχή έγινε στι 19 Φεβρουαρίου, τον περασμένο μήνα στην Άγκυρα και το Συμβούλιο θα συνεχίσει να υποστηρίζει την Επιτροπή στις προσπάθειές της να επιτύχει μια ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων όσο πιο θετική γίνεται. Επίσης θα ζητήσει την συνεργασία μεταξύ Frontex και Τουρκίας ο κανονισμός 207-2007 ε, ενισχύει αυτή τη μορφή συνεργασία με τρίτε χώρε. και πρέπει να σας πω επίσης ότι οι διαπραγματεύσεις για μια τέτοια συμφωνία όπως αυτή που προβλέπει ο κανονισμός μεταξύ Frontex και Τουρκίας συζητείται αυτή τη στιγμή. Έχουμε μπροστά μας μια επιχειρησιακή δραστηριότητα, ανταλλαγή πληροφοριών, ε, διαπίστωσης κινδύνου, ερευνητικές δραστηριότητες. Είναι ένα έργο κοινών συντονισμένων δράσεων του Frontex. Αυτό είναι το πλαίσιο μέσα στο οποίο εξελίσσεται η επιχειρησιακή συνεργασία μεταξύ της υπηρεσίας Frontex και των τουρκικών αρχών. Ελπίζουμε ότι οι διαπραγματεύσεις αυτές θα τελειώσουν το συντομότερο δυνατό με καρποφόρα αποτελέσματα και ούτως ή άλλως θα συνεχίσουμε να, σας, να ενημερώνουμε τα κράτη-μέλη για όλες τις εξελίξεις που θα λάβουν χώρα στο εγγυς μέλλον. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σίγουρα έχετε συμπληρωματική ερώτηση κύριε Παπα-Νικολάου. Μικρόφωνο σας ευχαριστώ πολύ για την απάντησή σας. θα ήθελα να συνεχίσω με δύο ακόμη σχόλια. το πρώτο είναι ότι σήμερα ή αύριο παράλληλα με τη συζήτηση που έχουμε σήμερα στην ελληνική βουλή ε, ψηφίζεται νομοθετική πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης η οποία καθιστά πιο ελαστική και πιο εύκολη την απόκτηση ελληνικής ηθαγένειας σε σχέση με το παρελθόν και βεβαίως αυτό καθιστά την ελλάδα ακόμη πιο μεγάλο πόλο έλξης για του μετανάστε, γιατί πιστεύουν μελλοντικά βεβαίω, ειδικά οι παράνομοι ότι κάποια στιγμή θα μπορέσουν να νομιμοποιηθούν. θα ήθελα από στρατηγική απόψεως την τοποθέτηση τη Προεδρία για το κατά πόσο αυτό είναι σωστό. και δεύτερο ε, ε, ανακοινώθηκε το φεβρουάριο ότι η frontex θα δημιουργήσει παράρτημα το πρώτο της παράρτημα στον πειραιά για την ενδυνάμωση της παρουσίας στο αιγαίο. αν γι' αυτό έχουμε ε, κάποιο πιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. σας ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, κύριε Βουλευτά, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να σας δώσω συγκεκριμένα στοιχεία για το χρονοδιάγραμμα των διαπραγματεύσεων αυτών. Είναι βέβαιο ότι υπάρχει πολιτική βούληση για το σκοπό αυτό τα στοιχεία που μας είπατε, το γεγονός που μας αναφέρατε για την Ελλάδα, αυτό που τονεί, που εμφανίζει ως ε, πρόδειλο είναι ότι η ανάγκη της καταπολέμησης της παράνομης μετανάστευσης να ενισχυθεί μέσω αυτών των συμφωνιών επανεισδοχής. Εμείς πρέπει να υποστηρίξουμε τις συζητήσεις που διεξάγει κατά βάση η Επιτροπή Πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι ήδη πριν το τέλος του, έτ, του περασμένου έτους υπήρξε μια επίσκεψη της Υπουργού κυρίας Μπίλστρομ ε, από την Σουηδική Προεδρία και του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Μπαρός στην Τουρκία, 5 Νοεμβρίου συγκεκριμένα, που ακολουθήθηκε από επαφές της Επιτροπής, της νέας πλέον Επιτροπής, που σε αυτή την περίπτωση θα αποτελεί αρμοδιότητα της κυρίας Μάλστρον που γνωρίζει πολύ καλά το πρόγραμμα της Στοκόλμης διότι μετέσχε στην προετοιμασία και την υλοποίησή του. Είμαι κατά συνέπεια αισιόδοξο ότι αυτά τα γεγονότα που αναφέρετε θα καλυφθούν, θα αντισταθμιστούν από μια ισχυρότερη, πολύ ισχυρότερη ρύθμιση των συμφωνιών επανεισδοχής, τη δημιουργία ουσιαστικά τέτοιων συμφωνιών επανεισδοχής με την Τουρκία. Ε, δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για αυτές τις συμφωνίες αυτή τη στιγμή. Μπορώ να σας βεβαιώσω ωστόσο ότι η Προεδρία είναι αποφα... του Συμβουλίου αλλά και η Επιτροπή είναι αποφασισμένη να επιτύχουν αυτή τη συμφωνία επανεισδοχής με την Τουρκία. Όχι μόνο με την Τουρκία και με άλλες χώρες ε, από όπου είτε προέρχονται είτε περνούν παράνομοι μετανάστες. Να σας πω επίσης ότι οι συμφωνίες της Frontex στη συγκεκριμένη περίπτωση με την Τουρκία διεξάγονται απευθείας από την ίδια την Frontex. Είναι συζητήσεις με τεχνικό και επιχειρηματικό χαρακτήρα πολλές από αυτές και το Συμβούλιο ναι μεν δεν εμπλέκεται στις διαπραγματεύσεις αυτές, ωστόσο ενημερώνεται και βεβαίως το Συμβούλιο θα ενημερώσει τα υπόλοιπα κράτη-μέλη και την Ελλάδα, όπως είναι αυτονόητο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Μια συμπληρωματική ερώτηση από τον κύριο Φάνσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι γίνονται συνομιλίες μεταξύ Frontex και Τουρκίας και για αυτές τις συνομιλίες ενημερώνεται η Επιτροπή, ενημερώνεται το Συμβούλιο. Θα ήθελα λοιπόν να μας ενημερώσετε να γνωρίζω αν η βάση αυτών των συζητήσεων μεταξύ τουρκίας και frontex γίνεται με βάση το σεβασμό των συνόρων ελλάδας τουρκίας δηλαδή με βάση την αναγνώριση και το σεβασμό των εξωτερικών συνόρων της τουρκίας. θυμίζω ότι μέχρι τώρα παρενόχληση των πτυτικών μέσων της frontex από την πλευρά της τουρκίας γινόταν με βάση αυτή την αμφισβήτηση και επίσης αν θέτει κάποιους άλλους όρους η τουρκία προκειμένου να συμφωνήσει με τη frontex. Προτού απαντήσετε κύριε Υπουργέ, υπάρχει από τον κύριο Χέλμα μια συμπληρωματική ερώτηση. Θέλω να συγχαρώ τον Υπουργό για τη θαυμάσια απάντησή του και την πολύ καλή δουλειά που κάνει την προστασία των δικαιωμάτων των μεταναστών. Ανησυχώ ότι κάποιε φορέ δεν προστατεύουμε τα δικαιώματα των δικών μα πολιτών που μετακινούνται από μία χώρα στην άλλη και αναφέρομαι στους ψηφοφόρους των Midlands οι οποίοι έχουν ξοδεύσει χρήματα για να αγοράσουν μια κατοικία στην Ισπανία για να διαπιστώσουν μετά από τρία χρόνια παραμονής ότι έφτασαν οι βουλντόζες στην πόρτα τους και ότι και η προσφυγή τους στην, στην δικαιοσύνη την Ισπανική αγνοήθηκε παντελώς. Ελπίζω λοιπόν να φροντίζετε καλύτερα για το, τις συνθήκες από τις οποίες ζουν οι πολίτες άλλων χωρών στην Ισπανία. Αφορούσε βεβαίως η ερώτηση μόνο την Τουρκία, αλλά θα επιτρέψω παρόλα τα αυτό στον Υπουργό να απαντήσει και στη δική σας ερώτηση. Κύριε Πρόεδρε, σε ό,τι αφορά την ερώτηση για την Ελλάδα, προφανώς πρόκειται για συμφωνίες οι οποίες περιλαμβάνουν σεβασμό των συνόρων των χωρών μερών της Ένωσης. Στις συμφωνίες αυτές ο στόχος ακριβώς είναι να υπάρξει σεβασμός των συνόρων. Όταν υπάρχει μια συμφωνία με μια τρίτη χώρα, μέσω της οποίας μπορεί να περάσει παράνομη μετανάστευση και υπάρξει συμφωνία επανεισδοχής, αυτός είναι ο στόχος. Άρα ενισχύονται οι συμφωνίες της Ένωσης με την τρίτη αυτή χώρα, φιλοσοφία της γενικότερης σφαιρικής έμφασης και του Συμφώνου για την Μετανάστευση και το Άσυλο είναι η ενίσχυση των συνόρων των χωρών μελών της Ένωσης. Αυτό είναι το αποτέλεσμα, η συνέπεια. Εάν δεν υπάρξει αυτή η αποτελεσματικότητα σε ό,τι αφορά τον έλεγχο τη παράνομη μετανάστευση, διότι δεν υπάρχει επαρκή συνεργασία από πλευρά τρίτων χωρών ή διότι δεν υπάρχουν συμφωνίε επανεισδοχή, αποδυναμώνεται στην πράξη το σύνορο αποδυναμώνονται ε, τα, τα όρια. Ο στόχος των διαπραγματεύσεων αυτών και οι συμφωνίες επανεισδοχής είναι η ενίσχυση των συνόρων, προφανώς και της Ελλάδος. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση του Βρετανού βουλευτή για τους Βρετανούς πολίτες που πήγαν στην Ισπανία, αγόρασαν, ε, επένδυσαν τις αποταμιεύσεις τους στην Ισπανία. Προφανώς εγώ δεν εκπροσωπώ την Ισπανία ως χώρα στις νομικές διαφορές που υπάρχουν με πολίτες ε, που βρίσκονται εκεί. Τα προβλήματα αυτά λύνονται σε ανεξάρτητα δικαστήρια. Εκπροσωπώ εδώ το Συμβούλιο της Ένωσης. Κατά συνέπεια δεν θα ήθελα να μιλήσω εξ ονόματος μιας συγκεκριμένης χώρας για συγκεκριμένα ζητήματα που δεν έχουν σχέση με, την με το Ευρωπαϊκό Δίκαιο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Υπουργέ. Περνάμε στην επόμενη ερώτηση της κυρίας Χάρκιν που αναφορά την ενδοοικογενειακή βία. Έχετε το λόγο. Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. Είναι γνωστό ότι η Ισπανική Προεδρία του Συμβουλίου της Ένωσης περιλαμβάνει μεταξύ των προτεραιοτήτων της την μάχη κατά της βίας κατά των γυναικών. Την ισότητα δηλαδή μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κάτι που δεν έχει επιτευχθεί 50 χρόνια μετά την γέννηση της Ένωσης. Ιδίως δε για την καταπολέμηση της μίζωνος διάκρισης, του μεγαλή, της μεγαλύτερης μάστιγας στην Ευρώπη και, στο, και σε όλες τις κοινωνίες του κόσμου, που είναι συγκεκριμένα η μάχη κατά της βίας κατά των γυναικών. Πρόκειται για έναν βασικό στόχο της Προεδρίας, διότι θεωρούμε ότι είναι ουσιώδης στόχος της Ευρώπης. Και για τον λόγο αυτό, επειδή ακριβώ είναι ένα στόχος της Ευρώπης, ένα πρόβλημα ευρωπαϊκών διαστάσεων, απαιτεί και μια ευρωπαϊκή επίση στρατηγική για την καταπολέμηση του φαινομένου αυτού. Και αυτό συνεπεριέλαβε στο πρόγραμμά τη η Ισπανική Προεδρία. Και όχι μόνο η Ισπανική Προεδρία και η Προεδρία του Τρίου με το Βέλγιο και την Ουγγαρία για το 18μηνο πρόγραμμα των Προεδριών. Είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που διότι το Κοινοβούλιο ήταν πάντα ένα όργανο που ήταν δραστήριο στον τομέα αυτό και συχνότατα απίφθινε εκκλήσεις προς την κατεύθυνση αυτή κατά της βίας, της έμφυλης βίας. Σε ένα ψήφισμα του περασμένου έτους ε, το Κοινοβούλιο ζήτησε από την Επιτροπή να επεξεργαστεί μια οδηγία, γενική οδηγία για μέτρα πρόληψης και καταπολέμησης όλων των μορφών έμφυλης βίας. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παρότρινε τα κράτη-μέλη να εξετάσουν ε, ε, διεξοδικότερα τις στατιστικές για την έμφυλη βία. Και ε, η Ισπανική Προεδρία ακριβώ βάσει αυτών των αιτήματων του Κοινοβουλίου θεώρησε την βία κατά τον γυναικών ως ένα ζήτημα κρίσιμο. Πιο συγκεκριμένα θεωρούμε ότι δημιουργεί δημιουργία παρατηρίου για την ενδοοικογενειακή βία, για την, βία, για την έμφυλη βία, συγγνώμη, κάτι που ξεκίνησε από το Συμβούλιο ΕΠΣΚΟ που υιοθέτησε στις 8 Μαρτίου, την περασμένη Δευτέρα δηλαδή, μια σχετική, ένα κάτι σχετικά συμπεράσματα, αλλά και την οδηγία για το ένταλμα προστασίας κατά της έμφυλης βίας. Πρόκειται για δύο ε, πολύ σημαντικές θεμελιώδεις πρωτοβουλίες που ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να εξελιχθούν και να ολοκληρωθούν πριν ολοκληρωθεί η εξάμεινη προεδρία της ε, Ισπανίας. Ευχαριστώ κυρία Χάρκιν, ευχαριστώ η Υπουργέ και θέλω να συγχαρώ την Ισπανική Προεδρία γιατί έδωσε τόση σημασία στην ε, ενδοοικογενειακή βία. Και πιστεύω ότι η πρωτοβουλία σας θα συνειδητοποιήσει και θα ευαισθητοποιήσει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. το ψήφισμα του Νοεμβρίου, στο ψήφισμα του Νοεμβρίου ζητεί το η δυνατότητα να υπάρξει μια σαφής νομική βάση για το θέμα αυτό. Θα υποστηρίξετε λοιπόν τις προσπάθειες της Επιτροπής για τη σύνταξη μιας ολοκληρωμένης, ολοκληρωμένης εμπεριστατωμένης έκθεσης για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας. Bueno, señora Κυρία Χάρκιν, κυρία Πρόεδρε, η συνθήκη της Λισαβόνας, όπως ξέρετε, θεσπίζει αλλαγή, επιφέρει μάλλον αλλαγή στη νομική βάση του ευρωπαϊκού δικαίου και στους κανονισμούς και στους οδηγίες, διότι ενσωματώνει στο λεγόμενο κοινοτικό πυλώνα τρεις διαφορετικούς πυλώνες. Την, τον κοινοτικό πυλώνα, τον πυλώνα της ΚΕΠΑ και τον πυλώνα της δικαιοσύνης και εσωτερικών υποθέσεων. Ενσωματώθηκαν όλα, όλα αυτά σε έναν πυλώνα, σε μία νομική προσωπικότητα και αυτό σημαίνει ότι και στον τομέα της εξωτερικής πολιτικής, ειδικότερα δε των θεμάτων δικαιοσύνης για την περίπτωση που μας αφορά, αστυνομική συνεργασία, ποινική και ε, αστική δικαστική συνεργασία, υπάρχει εισαγωγή της κοινοτική μεθόδου, της παραδοσιακή μορφής κοινοτική συνεργασίας, δηλαδή μεγαλύτερη παρουσία της επιτροπή, μεγαλύτερη παρουσία και του Κοινοβουλίου και δικαίωμα ελέγχου από το ΔΕΚ. Στον τομέα της ποινική συνεργασίας υπάρχει ακόμα μία εκκρεμότητα. Το 1 τέταρτο των κυβερνήσεων της Ένωσης μπορεί να αναλάβουν σχετική πρωτοβουλία. Αυτό συμβαίνει με το θέμα της οδηγίας για την έμφυλη βία. 12 κυβερνήσει, 12 κράτη υπέβαλαν πρωτοβουλία που εν τέλει πρέπει να αποφασίσει το Συμβούλιο και η Οδηγία γιατί αποτελούν θέματα της συναπόφασης. Οδηγία έλεγα η οποία βρίσκεται υπό διαπραγμάτευση τηρεί τις προϋποθέσεις της συνθήκης που επιτρέπει στις κυβερνήσεις να προχωρούν ε, σε νομοθετική πρωτοβουλία και σωστά νομίζω γιατί πρόκειται για, ποινική, ε, για συνεργασία στον τομέα της ποινικής δικαιοσύνης για αδικήματα ε, διότι η βία κατά ενός ατόμου οι σωματικές βλάβες κατά ενός ατόμου είναι αδίκημα κατά συνέπεια στόχος είναι η προστασία των θυμάτων της εγκληματική πράξη. Αυτή είναι η νομική βάση ποινική δικαστική συνεργασία. Ε, θεωρούμε ότι είναι σωστή και, το, ε, και η νομική υπηρεσία του Συμβουλίου ήδη γνωμοδότησε ότι μπορεί να προχωρήσει στη συζήτηση και να φτάσει εδώ πέρα. Ελπίζω, εδώ στην αίθουσα αυτή, ελπίζω ότι αυτό θα προχωρήσει γρήγορα γιατί ε, πρόκειται για ένα νομοθετικό κείμενο που το προσμένουν με ανυπομονησία εκατομμύρια ανθρώπων, γυναικών και ανδρών, πρέπει η καταπολέμηση της βίας να φύγει από την κρεβατοκάμερα και να μπει στην ευρωπαϊκή αρένα, στην ευρωπαϊκή διάσταση και να αποτελέσει αντικείμενο μέρημνα των κυβερνήσεων της Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν πολλές συμπληρωματικές ερωτήσεις. Θα δεχθώ μία από τον κύριο Μάρτιν και από τον κύριο Λότσεμ. Κύριε Μάρτιν πρώτος, ο κύριος Μάρτιν πρώτος. Ευχαριστώ πρόεδρε. Θα, όπως και η κυρία Χάρκιν συγχαίρω και εγώ την Ισπανική Προεδρία που έβαλε στην κορυφή της ατζέντα την ενδοοικογενειακή βία. Θέλω να αναφερθώ σε μία εμπειρία πριν από 20 χρόνια στο Εδιμβούργο έγινε μια εκστρατεία μηδενικής ανοχής και το συμπέρασμα της εκστρατείας και της έρευνας ήταν ότι χρειάζεται ευρύτερη ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων μερών. Η Κομισιόν ε, ε, έχει το Συμβούλιο θα σκεφτεί να εξετάσει αυτή την έρευνα και αυτή την έκθεση για να λύσει ενδεχομένω ορισμένα διδάγματα. Η βία δεν αφορά μόνο τις γυναίκες, αλλά δυστυχώς στρέφεται και κατά των παιδιών και πολλές φορές υπάρχει και ενδοοικογενειακή βία. Αυτή λοιπόν η ενδοοικογενειακή βία ε, θα ληφθεί υπόψη ε, κυρίως σε σχέση με το παρατηρητήριο, το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο, το οποίο πρόκειται να συσταθεί. Κύριε Υπουργέ, όταν είστε έτοιμος, παρακαλώ να απαντήσετε. Κύριε Μάρτιν, προφανώς η φιλοσοφία που διέπει την πρωτοβουλία που υποστηρίζει και το Κοινοβούλιο για την μάχη δια της νομίμου οδού της πιο αποτελεσματικής νόμιμης οδού του, της δικαστικής οδού που είναι βάση του κράτους δικαίου είναι η φιλοσοφία που θα μπορούσαμε να την αποκαλέσουμε μηδενική ανοχή στην βία κατά των γυναικών. Η στάση αυτή σχετίζεται με μια εικόνα της έμφυλης βίας με κάτι που εδώ και αιώνες εμπεριέχεται εν υπάρχει στην κοινωνική δομή των κοινωνιών μας. Άρα πρέπει να δώσουμε μία ολοκληρωμένη, σφαιρική ε, έμφαση στη μάχη κατά της έμφυλης βίας, ούτως ώστε να αποκτήσει αποτελεσματικότητα. Διότι είναι μια βία που πολύ δύσκολα μπορούμε να ξεριζώσουμε. Είναι βαθιά ριζωμένη και δύσκολα μπορεί να ξεριζωθεί. Για το λόγο αυτό και παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε εθνικό επίπεδο, συνεχίζουμε να υφιστάμεθα αυτή τη μάστιγα που σημαίνει και σε πολλές περιπτώσεις εμφανίζεται σαν την άκρη του παγόβουνου. Ε, το ποσοστό της βίας που γνωρίζουμε είναι ένα μικρό ποσοστό της πραγματικής ενδοοικογενειακής βίας. Άρα χρειάζεται να υπάρχει μια πλήρης συνεκτική αντιμετώπιση του ζητήματος χρησιμοποιώντας όλα τα νομικά εφόδια που έχουμε στη διάθεσή μας, ε, δημιουργώντας επίγνωση στα μέσα ενημέρωσης, μετα... ενσωματώνοντας την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού και στην... στο εκπαιδευτικό σύστημα. Και γι' αυτό μιλούσα και για την... το Συμβούλιο Κοινωνικών Υποθέσεων του... της Δευτέρας ε, που υιοθετήθηκε αυτή η προσέγγιση, μηδενική δηλαδή ανοχή της βίας κατά των γυναικών. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση του άλλου βουλευτού για την επέκταση της οδηγίας στη βία κατά των ε, παιδιών, ε, των ηλικιωμένων, βεβαίως πρόκειται για μια βία που ασκείται έναντι των περισσότερο ευάλωτων ανθρώπων. Το μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό, λένε σε πολλές χώρες μας. Στη χώρα μου τουλάχιστον. Η, στάση αυτή εμφανίζεται στην συγκεκριμένη μορφή βίας που έχει να κάνει με το πόσο ευάλωτος είναι το θύμα. Ο άνθρωπος που είναι πιο αδύναμος και δείχνει την δηλία αυτού που ασκεί τη βία στον πιο ευάλωτο. Τη γυναίκα, το παιδί, τον ηλικιωμένο. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που ε, ε, που, που, κάτω, πάνω στο οποίο στηρίζεται η όλη προσέγγιση. Γι' αυτό ζητούμε από την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα να υιοθετήσει την πρωτοβουλία ενός ευρωπαϊκού έτους ε, κατά της βίας ενάντια στις γυναίκες, στους ηλικιωμένους, στα παιδιά. Αυτό περιλαμβάνεται στο λεγόμενο πρόγραμμα Δάφνη 3 και δείχνει, κύριε Βουλευτά, ότι είναι αναγκαίο η προστασία αυτή να επεκταθεί σε όλες τις τρωτές ομάδες ανθρώπων. Παιδιά και ανηλίκους, για παράδειγμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Περνάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση που έχει υποβληθεί από τον κύριο Πόσελτ και αφορά τη στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη. Ευχαριστώ κύριε Πόσελτ. Η στρατηγική για το Δούναβι είναι ένα από τα θέματα που εξετάζει το πρόγραμμα του τρίου προεδριών Ισπανίας, Βελγίου, Ουγγαρίας. Όπως φαντάζεστε μετά από πρωτοβουλία της Ουγγαρίας. Υιοθετήθηκε η στρατηγική αυτή για το Δούναβι. Οι τρεις λοιπόν χώρες έχουμε δεσμευθεί να προχωρήσουμε αυτή τη στρατηγική για την λεκάνη του Δούναβη και το Συμβούλιο παρότρινε πέρυσι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, συγγνώμη, ε, παρότρινε πέρυσι την Κομισιόν να υποβάλει το σχέδιο στρατηγική για το Δούναβη πριν τελειώσει το έτο. Περιμένουμε την ε, υποβολή του σχετικού σχεδίου από πλευρά τη Επιτροπή. Η Επιτροπή αυτό που έκανε ήταν να ξεκινήσει μία δημόσια διαβούλευση η οποία θα κρατήσει μέχρι τον Μάρτιο φέτος και μετά βάσει των αποτελεσμάτων της δημόσιας διαβούλευσης η Επιτροπή θα προτείνει την στρατηγική που ελπίζουμε να υιοθετηθεί επίσημα ε, τον Δεκέμβριο του φετινού έτους μετά από μια ανακοίνωση της Επιτροπής. Περιμένουμε την ανακοίνωση αυτή. Θέλω ωστόσο να σας ε, ενημερώσω ότι έλαβε χώρα μια σημαντική συνάντηση στην οποία υπήρξε σημαντική πρόοδος για την εξέλιξη στρατηγικής αυτής στις 25 ε, Φεβρουαρίου τον περασμένο μήνα δηλαδή στη Βουδαπέστη με εκπροσώπους ε, των κυβερνήσεων της Αυστρίας, της Βουλγαρίας, της Τσεχίας, της Γερμανίας, της Ουγγαρίας, της Ρουμανίας, της Σλοβακίας, της Σλοβενίας Συνάντηση η οποία υιοθέτησε μια σειρά σημαντικών συμπερασμάτων για τα βασικά στοιχεία αυτής της μελλοντικής στρατηγικής. Όπου στόχος είναι η θέση από κοινού, η από κοινού εκμετάλλευση των πόρων και των δυνατοτήτων που έχουν οι χώρες αυτές χρησιμοποιώντας με έναν οικονομικά ουδέτερο τρόπο ευρωπαϊκούς πόρους ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι προόδου κοινωνικής, οικονομικής και τουριστικής ανάπτυξης ενός κάποιου μεγέθους. Περιμένουμε, όπως σας είπα, την ανακοίνωση της Επιτροπής για το θέμα αυτό, που θα ξεκινήσει όταν ολοκληρωθεί η δημόσια διαβούλευση. Κατόπιν το Συμβούλιο όταν έχει την ανακοίνωση στα χέρια της θα ε, προχωρήσει στην αξιολόγησή της. Σίγουρα έχετε συμπληρωματική ερώτηση κύριε Πόσετ. παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για την διεξοδική επάνηση. Μόνο μία σύντομη ερώτηση. Αυτή η στρατηγική του Δούναβη αφορά τις μεταφορές και τον πολιτισμό. Θεωρώ ότι και οι δύο είναι πολύ σημαντικοί για τη διασυνοριακή συνεργασία. Και θέλω να ερωτήσω κατά πόσον υπάρχει ε, οριστικός κατάλογος ε, των κρατών που θα συμπεριλαμβάνονται ή κατά πόσον αυτό ακόμα πρόκειται να αποφασιστεί. Γιατί το Κοινοβούλιο πρότεινε κάποια διεύρυνση του καταλόγου. Ο κύριος Υπουργό έχει το λόγο. Ε, δεν είναι η πρόεδρο του Συμβουλίου που θα αποφασίσει τον καταλόγο των χώρων. Το καταλαβαίνετε αυτό. Οι κυβερνήσει που σας ανέφερα θέλουν να προχωρήσουν με τη στρατηγική αυτή, ενδιαφέρονται να την αναπτύξουν και περιμένουν να γίνει η ανακοίνωση της Επιτροπής. Μπορώ να σας πω επίσης ότι οι εν λόγω χώρες θεωρούν πως η στρατηγική αυτή πρέπει να παίξει ρόλο πρωτοπορίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην Κομισιόν ιδιαίτερα, διευκολύνοντα την συνεργασία στην περιοχή του Δουνάβεως. Στην δήλωση που ανέφερα προηγουμένως στις 25 Φεβρουαρίου αναφέρεται ότι η στρατηγική για την περιοχή του Δουνάβεως πρέπει να χρησιμεύσει για να αυξηθεί η ευημερία, η ασφάλεια και η ειρήνη στους λαούς που ζουν στην περιοχή αυτή μέσω μιας διαπεριφερειακής και διεθνικής συνεργασίας και συντονισμού και να καλύψει στρατηγικούς τομείς πολιτικής όπως την ενέργεια, το περιβάλλον, την προστασία της φύσης, τις μεταφορές, τις υποδομές, την καινοτομία, τις πολιτιστικές και καλλιτεχνικές δραστηριότητες την βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, τον τουρισμό, την επισητιστική ασφάλεια, την οικονομία, την συνεργασία μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων, την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, την μετανάστευση, τον αθλητισμό, την εκπαίδευση, την υγεία, κοινωνικά ζητήματα και άλλες πτυχές που περιλαμβάνει με πολύ φιλόδοξο και διεξοδικό τρόπο το κείμενο αυτό, ένα πολύ σημαντικό κείμενο, που θεωρώ σκόπιμο, να αναφέρω λόγω της ερώτησης που θέσατε και για την οποία σας ευχαριστώ. Πιστεύω ότι πρόκειται για ένα φιλόδοξο στόχο. Περιμένουμε την διαβούλευση αυτή και την, ακίνηση και την των επιτροπής. Βεβαίως υπάρχει πάντως η πολιτική βούληση μεταξύ των τριών μελών του τρίου της Προεδρίας υπάρχει πολιτική βούληση για να προχωρήσει η στρατηγική αυτή για τον Δούναβη. Ευχαριστώ Κύριε Υπουργέ, υπάρχουν πολλές συμπληρωματικέ ερωτήσεις. Πρέπει να λάβουμε υπόψη τη σειρά με την οποία κατατέθηκαν αυτές οι ερωτήσεις και τις πολιτικές ομάδες από τις οποίες προέρχονται. Γι' αυτό θα δεχθώ τι ερωτήσει τις ερωτήσεις του κυρίου Ρούμπικ και Τικάου. Κύριος Ρούμπικ πρώτος. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Πρόεδρε, ο Δούναβης είναι ποταμός και στην περίπτωση του ποταμού πρέπει κανείς ε, να προσέχει και την καθαρότητά του. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό τι είδου εγκαταστάσει ε, καθαρισμού ε, υπάρχουν στον ποταμό για να βελτιώνεται η ποιότητα των νερών του ποταμού. Για μας ο στόχος είναι ο δούναβη να έχει πόσιμο νερό από την αρχή μέχρι το τέλος. Εσεί πιστεύετε ότι μπορεί ο Δούναβή να χρησιμοποιηθεί για την υδροηλεκτρική ενέργεια, την παραγωγή τη ή και για την αποθήκευση νερού έτσι ώστε στην Ευρώπη να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια όσον αφορά την ενέργεια. Ευχαριστώ κυρία Τικάου. Thank you, Madam Chair. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Δούναβι θα στηριχθεί σε ένα φιλόδοξο σχέδιο δράσης το οποίο να προσδιορίζει συγκεκριμένες προτάσεις και ενέργειες υπέρ των κατοίκων των χωρών μέσα από τις οποίες περνάει ο Δούναβης. Έχει ξεκινήσει η δουλειά για την υλοποίηση ενός τέτοιου σχεδίου και με βάση ποιων κριτηρίων θα γίνει η επιλογή των σχετικών έργων και προγραμμάτων. Έχετε το λόγο, κύριε Υπουργέ. Προφανώ ο στόχος που ανέφερε ο κύριος Ρούμπικ θα ε, συμπεριληφθεί στην στρατηγική του Γνάβερος. Εγώ μίλησα νωρίτερα για την, τις διαστάσεις της στρατηγικής αυτής και τους στόχους της, που είναι στόχοι σημαντικοί, καλύπτει ένα τεράστιο αριθμό ζήτηματων που επηρεάζουν τη ζωή των ανθρώπων που ζουν στην περιοχή, την καθημερινότητά τους, σχετίζονται με την οικονομία, τον πολιτισμό, την προστασία του περιβάλλοντος και τους φυσικούς πόρους μεταξύ των οποίων και το νερό προφανώς. αυτό το, αυτός ο φυσικός πόρος είναι αυτονόητος στην οτροπία της περιοχής και προφανώς θα συμπεριληφθεί, είμαι πεπισμένος, στην στρατηγική αυτή που κατά βάση, τις οποίες κατά βάση θα ηγηθούν οι χώρες που προωθούν την στρατηγική αυτή και που τις προανέφερα και που συναντήθηκαν πριν από λίγο, λίγες μέρες στην Βουδαπέστη για να προχωρήσουν στον ορισμό των στόχων την συγκεκριμενοποίηση της στρατηγικής που ακόμα δεν έχει οριστεί επαρκώς. Για το λόγο αυτό πιστεύω ότι είναι πρόημο να μιλούμε και μιλώ για την παρέμβαση της κυρίας Τικάου να ε, μιλάμε για κριτήρια επιλογής έργων ή επιλεξιμότητα έργων. Είναι πρόημο αυτό. Φαντάζομαι ότι θα σχετίζονται με το πόσο συναφή είναι τα έργα, με τους στόχους που προανέφερα. Αλλά μπορεί να προσθεθούν και άλλα κριτήρια και άλλα ζητήματα. Ναυσιπλοεία, ε, ενεργειακή ασφάλεια, ε, ανάπτυξη της υπαίθρου, δημογραφικά ζητήματα, μάχη κατά της αλλαγής του κλίματος, συνέπειες των αλλαγών των οικονομικών αγορών. Και άλλα ζητήματα που μπορεί να απασχολούν τους κατοίκους της περιοχής. Θέματα που απαιτούν παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που απαιτούν, που ενδιαφέρουν την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της και τις ουσιαστικές πολιτικές της. Είμαι πεπισμένος ότι όλα αυτά τα ζητήματα θα αποτελέσουν αντικείμενο της προσοχής των κρατών μελών. Η, η συνοχή, για παράδειγμα. Όχι μόνο η κοινωνική συνοχή, αλλά και ένα καινούριο στοιχείο της συνθήκης της Λισαβόνας που είναι η εδαφική συνοχή, που είναι μια νέα μορφή συνοχής που εμφανίζεται με τη συνθήκη της Λισαβόνας και σχετίζεται πολύ, ταιριάζει πολύ με αυτή την πρωτοβουλία για την στρατηγική για το Δούνευ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Περνάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση Πρόκειται, και θα συνδυάσουμε τις ερωτήσεις 4 και 5, την ερώτηση του κυρίου Πουπάκη δηλαδή για το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Μοντέλο και αντιμετώπιση Φτώχειας και την ερώτηση του κυρίου Έλβορντ για το Ευρωπαϊκό Έτος για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού για να σας καθησυχάσω και τους δύο θα έχετε τη δυνατότητα να υποβάλλετε συμπληρωματικές ερωτήσεις στον Υπουργό αφού μας δώσει μια κοινή απάντηση και για τις δύο ερωτήσεις. Uh, Είπατε δύο ερωτήσεις κυρία Πρόεδρε. Checked. Ακριβώς και σας, ε, μας είπαν ότι θα απαντήσετε και στις δύο ερωτήσεις ε, μαζί. Ευρωπαϊκό κοινωνικό μοντέλο για καταπολέμηση της φτώχειας. Αυτές είναι οι δύο ερωτήσεις. Κύριε Πρόεδρε, η Προεδρία συμμερίζεται την άποψη των κύριων βουλευτών για την ανάγκη να υπάρξει ψηλό επίπεδο κοινωνικής προστασίας, ιδίως των ομάδων που απειλούνται από φτώχεια και από κοινωνικό αποκλεισμό που αποτελεί ένα από, τον ακρογωνία, από λήθους του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου, ιδίω σε μια χρονική στιγμή κατά την οποία βρισκόμαστε σε περίοδο οικονομικής ε, ύφεση, ανεργίας. Η ανεργία υπολογίζεται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση των ανέργων κατά 5 εκατομμύρια σε σχέση με το ξεκίνημα της περίοδου της κρίσης. Είναι πολλοί αυτοί που εκτίθενται σε κίνδυνο φτώχειας ή υπερχρέωσης. Είναι πολύ πιθανό λοιπόν να συνεχίσουν για κάποιο χρόνο τα ποσοστά της ανεργίας να παραμένουν υψηλά. Άρα η μακροχρόνια ανεργία να αποτελέσει αιτία κοινωνικού αποκλεισμού. Οι κοινωνικές λοιπόν συνέπειες της οικονομικής κρίσης θα είναι ένα βασικό θέμα στην ευρωπαϊκή πολιτική ημερήσια διάταξη των επόμενων μηνών. σίγουρα είναι ένα θέμα που απασχολεί το τρίο. Όχι μόνο τη δική μας προεδρία. Έχουμε ένα εργαλείο για την αντιμετώπιση του προβλήματος αυτού που είναι η απόφαση να θεωρηθεί το έτος 2010 ως Ευρωπαϊκό έτος κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που έχει τέσσερις βασικούς στόχους την αναγνώριση της αξιοπρέπειας των ανθρώπων και του δικαιώματος να παίξουν έναν ε, ενεργό ρόλο στην ε, κοινωνία, τον δημόσιο ρόλο της αντιμετώπισης ε, του αποκλεισμού, την συνοχή της κοινωνίας και την χρησιμοποίηση όλων των επιπέδων διακυβέρνησης μακροπρόθεσμο επίπεδο, σε μακροχρόνιο επίπεδο για την αντιμετώπιση της φτώχειας. Θα μιλήσω για μια έννοια που χρησιμοποίησα σε μια προηγούμενη απάντησή μου την προστασία των πιο ευάλωτων, αυτών που υποφέρουν περισσότερο και με διπλό τρόπο από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Μιλώ για τα παιδιά, τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους. Εμείς λοιπόν θα υποστηρίξουμε τις διάφορες πρωτοβουλίες που μπορεί να ανακύψουν για την αντιμετώπιση της φτώχειας και του αποκλεισμού θα ήθελα να σας πω ότι αυτό ελπίζω ότι θα γίνει κεντρικός στόχος ολόκληρης της στρατηγικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας στην Ένωση. Γιατί είναι ένας από, ένας από τους πιο εύκολα ποσοτικοποιημένους ε, στόχους της Επιτροπής που παρουσίασε την περασμένη ε, στις 3 Μαρτίου είναι το η δυνατότητα να προστατεύσουν 20 εκατομμύρια ατόμων που βρίσκονται στα όρια της φτώχειας σήμερα. Ευχαριστώ. Θα δεχθούμε τις ε, συμπληρωματικές ερωτήσεις αρχίζοντας με τον κύριο Πουπάκη. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ για την απάντησή σας. Θα ήθελα όμως ε, με τα σημερινά δεδομένα την ανεργία που όπως είπατε και εσείς το 2009 αγγίζει το 10% και το 45% των Ευρωπαίων ανέργων να παραμένουν εκτός αγοράς εργασίας για παραπάνω από ένα χρόνο την άναρχη επέκταση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης με την έλλειψη σαφούς θεσμικού πλαισίου όλα αυτά έχοντας δημιουργήσει 19 εκατομμύρια φτωχούς ανέργους θα θέλαμε να ενημερωθούμε γιατί είστε συγκεκριμένος μέχρι σήμερα και χαίρομαι γι' αυτό ποια συγκεκριμένα άμεσα μέτρα ενεργητικές και παθητικές πολιτικές απασχόλησης πρόκειται να υιοθετήσετε σε ευρωπαϊκό επίπεδο έτσι ώστε να αντιμετωπιστεί ουσιαστικά το ζήτημα των φτωχών εργαζομένων και των ανέργων ειδικότερα των μακροχρόνιων ανέργων γιατί θα αντιμετωπίσουν πρόβλημα και άμεσης επιβίωσης ακόμα πάντα με μέτρα σύμφωνα με τις αρχές και το πνεύμα του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. ευχαριστώ. Mr. Elwood. Μπορεί να μας πει το Συμβούλιο πώς θα εξασφαλίσει ότι η σύσταση για την ε, συμπερίληψη και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού θα εφαρμοστεί και πώς θα ενταχθεί στη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020 ώστε να σημειωθούν πρόοδοι στις προσπάθειες καταπολέμησης και μείωσης της φτώχειας. Sí, señora Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να επαναλάβω ότι έχουμε μπροστά μας ένα πρόβλημα όπου για πρώτη φορά με τόσο φιλόδοξο τρόπο υπάρχει πρόθεση να διαμορφωθεί μια ευρωπαϊκή στρατηγική. Μιλώ για τη μόχη κατά της φτώχειας, του αποκλεισμού και την ενεργό ένταξη των ιδίως μακροχρόνιων έργων, των ατόμων σχετικά μεγάλης ηλικία και επανερχόμαστε σε αυτό που σας είπα νωρίτερα, των πιο ευάλωτων δηλαδή. Ξεκινώντας, η Ευρωπαϊκή Ένωση με την ευκαιρία της οικονομικής κρίσης που βιώνουμε ξεκίνησε μια συντονισμένη βραχυπολιτική, βραχυπρόθεσμη ε, στρατηγική σοκ θα τη λέγαμε ένταξη ε ε, ε, ε, ε, παροχής δημοσίων κονδυλίων στην ιδιωτική πρωτοβουλία για στόχους κοινωνικής προστασίας όπως προστασίας δηλαδή του κράτους πρόνοιας για να μπορέσουν να δημιουργήσουν μια αντίδραση που είχε συνέπειες έστω και επιφανειακές συνέπειες για τα άτομα εκείνα που βρισκόντουσαν σε μακρά ανεργία και που δύσκολα, βραχυπρόθεσμα τουλάχιστον, θα μπορούσαν να βρουν μια νέα θέση στην αγορά εργασία. Άρα υπήρξε μια αντίδραση που πρέπει να λάβουμε υπόψη γιατί είναι μια πραγματική, υφιστάμενη, άμεση, έστω βραχαίως αντικτύπου παρέμβαση της Ένωσης. Επιπλέον η Ένωση υιοθέτησε μια στρατηγική για την καταπολέμηση της φτώχειας που είναι αποτέλεσμα της ανεργίας μακράς διάρκειας, μακροχρόνιας ε, για κατάρτιση, εξειδίκευση ή ανακύκλωση επανε, ή για ολοκλήρωση μιας μη ολοκληρωθήσης ε, εκπαίδευσης όταν ήταν κάποιος νέος για να δημιουργήσουν προϋποθέσεις απασχολησιμότητας. Κάτι πολύ σημαντικό και περιλαμβάνεται στη στρατηγική του, 20, του 2020 που ανέφερα προηγουμένω και που συμπεριλαμβάνεται στα συμπεράσματα του Συμβουλίου Κοινωνικών Υποθέσεων που συχνά αναφέραμε σήμερα τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα 8 του μηνό. Μια ευρωπαϊκή στρατηγική που θα εντάσσεται στου βασικού στόχου τη Ένωση όπω είναι αυτοί που περιλαμβάνονται στην στρατηγική της Ευρώπης του 2020. Ένας από τους ε, ποσοτικομοιημένους αυτούς στόχους που θα δούμε αν θα εγκριθούν στις 25-26 στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα εξετάσει την ανακοίνωση της Επιτροπής και θα εγκρίνει τους ποσοτικοποιημένους αυτούς στόχους. Ένας από τους οποίους είναι η μείωση κατά 20% του αριθμού, του ποσοστού των ατόμων που βρίσκονται ε, σε κίνδυνο φτώχεια. Μην ξεχνάτε ότι στην Ευρώπη υπάρχουν 80 εκατομμύρια άτομα που κινδυνεύουν να, μπουν, να, να βρεθούν σε καθεστώ φτώχεια, προσπαθώντα να μειώσουν το στόχο αυτό και να αυξήσουν την ενεργή ε, δραστηριότητα των ατόμων αυτών σε βράχη, σε βράχη και μέσο πρόθεσμη προοπτική με συντονισμένο τρόπο. Το κλειδί, κύριε και κύριοι, είναι ο συντονισμός των πολιτικών απασχόλησης και των κοινωνικών πολιτικών. Το λέει ξεκάθαρα η συνθήκη τη Λισαβόνα. Χρειάζεται να υπάρξει συντονισμό των κοινωνικών πολιτικών, των πολιτικών απασχόληση. Και αυτό είναι αυτό που προσπαθεί, ξεκινά να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση η υπό το βάρος της κρίσης. Αυτό είναι μια σημαντική εξέλιξη από την κρίση ε, με βάση τα εργαλεία που διαθέτει η Ένωση όπως την εσωτερική αγορά και τα διαθροτικά ταμεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Ελπίζω να μην μπερδέψαμε τα πράγματα υποβα... Ε, παίρνοντας μαζί δύο ερωτήσεις. Υπάρχουν... Επειδή υπάρχουν δύο ερωτήσεις, όπως θα, θα, δεχθώ όπως θα έκανα και για μία ερώτηση, δύο σύνολα, δύο συμπληρωματικών ερωτήσεων. Οι πρώτες δύο συμπληρωματικές ερωτήσεις θα είναι της κυρίας Φόρντ και του κυρίου Κόζου. Η κυρία Φόρντ πρώτη. Ευχαριστώ. Η οικονομική κατάσταση διαφέρει από χώρα σε χώρα και ευχαριστώ που αναφερθήκατε στις συντάξεις. Μπορεί να ε, ε, παρακρατήσει τα κονδύλια των ε, διαρθρωτικών ταμείων η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εάν δεν τηρούν τα κράτη-μέλη τις υποχρεώσεις τους. Το Κοινοβούλιο και τι γίνεται και θα θέλαμε να γνωρίζουμε τι ακριβώς προβλέπεται να γίνεται με τους κατόχους ιδιοκτησιών στην Ισπανία οι οποίοι πλήττονται από, ε, από μια σειρά προβλημάτων. Köszönöm szépen a szót. Egyetlen kérdésem. Κύριε Πρόεδρε, έχω μία και μόνο ερώτηση. Υπάρχουν ε, δύο ομάδες ε, οι οποίες θίγονται κατά κύριο λόγο από την φτώχεια. Πρόκειται για τους μη εκπαιδευμένους ε, και τους ανάπηρους. Δυστυχώ, τα προβλήματα αυτών των ομάδων δεν αντιμετωπίζονται παρκώ. Η δική μου ερώτηση λοιπόν είναι η εξής. Το Συμβούλιο προβλέπει να ασχοληθεί με τα προβλήματα αυτών των δύο ομάδων. Αυτών των δύο ομάδων. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ. Bien, eh, la primera pregunta sobre... Για την πρώτη ερώτηση. Ευχαριστώ για τους ε, συνταξιούχους που είναι ιδιοκτήτη κινήτων στην Ισπανία. Ε, παρόμοια με μια προγενέστερη είναι. Η απάντηση θα είναι και αυτή παρόμοια με αυτήν που έδωσα προηγουμένω. Πρόκειται για ένα θέμα που αφορά την εφαρμογή εσωτερικού νόμου ενός κράτους μέλους. Η εφαρμογή του ε, αυτή είναι, εγώ δεν μπορώ να μιλήσω για το θέμα αυτό εξ του Συμβουλίου που έχει την έξοδο στην δικαστική οδό, στην, ε, στην εθνική δικαστική οδό. Αυτό γίνεται παντού και πάντα. Για την ερώτησή σας σχετικά με τις ευάλωτες ομάδες, συμφωνώ απόλυτα με το να δώσουμε συγκεκριμένη και ειδική έμφαση στις δύο αυτές κατηγορίες που ανέφερε η κυρία Βουλευτής. Επιπλέον, διότι βρισκόμαστε σε μια χρονική στιγμή που έχουμε ένα νέο εργαλείο που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, τον χάρτη των θεμελιωδών δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που μιλά για τα δικαιώματα των ιδιαίτερα ευάλωτων ομάδων, ηλικιωμένοι, άτομα με αναπηρίες, και την ανάγκη προστασίας τη αξιοπρέπεια τους, αλλά και το δικαίωμα συμμετοχής του στην κοινωνική και πολιτιστική ζωή, αλλά ε, ευρύτερα στην προστασία τη αξιοπρέπεια της ε, σωματικής και ψυχικής ακεραιότητάς τους από απάνθρωπες ή εξεφελιστική, από απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση. Η εξευτελιστικη απο απανθρωπη Ένωση έχει διαμορφώσει μια σειρά εργαλείων και μέσων για την καταπολέμηση της κατάστασης αυτής Μεταξύ αυτών ασχολήθηκε ιδιαίτερα με την κατάστασή τους και μια μελέτη του Ευρωβαρομέτρου του 2007 είναι πολύ ενδιαφέρουσα γιατί το ίμιση των Ευρωπαίων, λέει το Ευρωβαρόμετρο του 2007, θεωρεί ότι οι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν κακή συμπεριφορά και κατάχρηση ακόμα όταν προσπαθούν να εκμεταλλευτούν, να, να απαιτήσουν τα δικαιώματά τους. Και αυτό το σκέφτεται το ίμιση των Ευρωπαίων. Δηλαδή, οι μισοί Ευρωπαίοι θεωρούν ότι η κοινωνία αντιμετωπίζει άσχημα τους ηλικιωμένους. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνεχίζει τη λεγόμενη ανοιχτή μέθοδο συντονισμού στον τομέα αυτό μεταξύ των κρατών μελών για τα ζητήματα κοινωνικής προστασίας. Θέλω να σας πω ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουμε μπροστά μας θέματα που στηρίζονται ε, ή που έχουν ε, εθνική διάσταση, που είναι, ανήκουν στην εθνική αρμοδιότητα, άρα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τα κράτη-μέλη, ιδίω με βάση την εφαρμογή τη αρχή τη επικουρικότητα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να συνοδεύσει τι πολιτικέ αυτέ, δεν μπορεί να τι υποκαταστήσει, καθόλου μάλιστα. Μπορεί να τι ε, συνοδεύσει, να τι επικουρήσει. Η κοινωνική διάσταση ωστόσο τη δημιουργία ε, θέσεων εργασία αναδεικνύεται σημαντικά στο τελευταίο αυτό κείμενο τη Επιτροπή και θα συζητηθεί στα τέλη Μαρτίου από του αρχηγού και και κυβερνήσεων. Η κοινωνική αυτή διάσταση θα πρέπει να εστιάζει την προσοχή τη στα ζητήματα που αναφέρθηκαν, χωρί να αγνοείται η προγενέστερη στρατηγική. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μα προφανώ τον κοινωνικό αντίκτυπο τη κρίσης, γιατί αυτό είναι ο σημαντικότερο. Ευχαριστώ. Όπως σας είπα, θα επιτρέψω και άλλες δύο συμπληρωματικές ερωτήσεις για το κοινωνικό μοντέλο και την καταπολέμηση της φτώχειας. Άτκινς και Χάνον. Κύριε Άτκινς πρώτα. τι πρόκειται να κάνει ο Υπουργό που εκπροσωπεί το Συμβούλιο για να προστατεύσει άτομα που απειλούνται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό σαν αποτέλεσμα τη πολιτική τη Ισπανία σε κατοίκου, σε υπηκόου Βρετανού και άλλων χωρών, των οποίων απαλωτριώνονται οι περιουσίε. Ο Υπουργό εξ ονόματο τη Προεδρία δεν μπορεί να αποφύγει το θέμα. Πρέπει να καλέσει την Ισπανική κυβέρνηση να λάβει τα αναγκαία μέτρα ο κύριος Χάνων και σας θυμίζω ότι το θέμα, ε, ε, το ποιο είναι το θέμα της ερώτησης που αυτή τη στιγμή εξετάζουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με τη φτώχεια των Ευρωπαίων πολιτών που βρίσκονται σε τμήματα της Ισπανίας. Καταλαβαίνω ότι είστε εδώ ως εκπρόσωπος Τη εκτελεστική εξουσία, όχι τη δικαστική ε, εξουσία τη Ισπανία. Δεν μπορεί να, να εκπροσωπείται μάλιστα την ε, κοινότητα τη Βαλένθια, την αυτόνομη περιφέρεια τη Βαλένθια. Υπάρχουν ωστόσο καταχρήσει που δεν έχουν να κάνουν με, την, με το νόμο αλλά με την εφαρμογή του νόμου. Αυτό είναι κάτι που μπορεί να επιληθεί. Ζήτω απλά να υπάρξει μια έρευνα της Ισπανικής κυβέρνησης για συγκεκριμένες καταχρήσεις. Είναι εντυπωσιακά τα ισπανικά σα, κύριε Χάνοκ, αλλά βεβαίω θα αποφασίσει ο υπουργό αν θέλει να απαντήσει ή όχι. Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να καταχραστώ τι θέσει μου ω Προεδρεύοντος του Συμβουλίου για να υποστηρίξω μια συγκεκριμένη κυβέρνηση ή ένα συγκεκριμένο εθνικό νόμο. Δεν θέλω να καταχραστώ τι θέσει μου αυτή, διότι σίγουρα θα με κατηγορούσαν ότι χρησιμοποιώ το βήμα αυτό για να, για να υποστηρίξω τις ε, δράσει συγκεκριμένη κυβέρνηση συγκεκριμένων χωρών. Ξέρετε πολύ καλά ότι το θέμα αυτό είναι ένα θέμα που αφορά, είναι καθαρά εθνικό. Έχει λύση σε εθνικό πλαίσιο. Και όχι μόνο η Ισπανία, αλλά και οι ευρωπαϊκές χώρες, όλες και οι 27, είναι χώρες που εφαρμόζουν κράτος δικαίου. Έχουν την κατάλληλη δικαστική οδό για να τάμουν τέτοιες περιπτώσεις πιθανών ε, ε, υποθετικών καταχρήσεων. Υπάρχει μια τέτοια οδός σε κάθε χώρα της Ένωσης. Και δεν μιλώ μόνο για την περίπτωση της Ισπανίας. Αυτό που συμβαίνει ή φαίνεται ότι συμβαίνει αντίστοιχα σε άλλες, ε, σε χώρες. Μπορεί και αλλού να υπάρχουν, όπου πάνω, θεωρείται ότι υπάρχει κατάχρηση, υπάρχει και, δια, και οδός. Αυτό σημαίνει όπου και να γίνεται. Είναι προφανές ότι το θέμα αυτό δεν είναι θέμα που δεν θέλω, για το οποίο θέλω, να, το οποίο θέλω να, ε, από το οποίο θέλω να υπεκφύγω. Καλά κάνετε εσεί και χρησιμοποιείτε το κοινοβούλιο για να παρουσιάσετε τι θέσει σα. Εγώ δεν θέλω να χρησιμοποιήσω το κοινοβούλιο για να απαντήσω σε ένα θέμα που είναι εσωτερικό ενό κράτου μέλου. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Περνάμε τώρα στην ερώτηση 6. Η ερώτηση 6 του κυρίου Χίγκιν αποσύρθηκε. Οπότε θα προσπαθήσουμε να συνδυάσουμε δύο ερωτήσεις, την 7 και την 8. 7 του κυρίου Παλέκης τον οποίο αντικαθιστά ο κύριο Πάντα απόψε με θέμα το καθεστώ των θεωρήσεων μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και της Ρωσίας η ερώτηση 8 ε, της κυρίας Αντρικένε που θα αντικατασταθεί απόψε από τον κύριο Πόσελτ με, θέμα σχέση Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας η ατζέντα της Ισπανικής Προεδρίας. Παρακαλούμε κύριε Υπουργέ να προσπαθήσετε να απαντήσετε σε συνδυασμό και στις δύο αυτές ερωτήσει. Κυρία Πρόεδρε, αν κατάλαβα καλά θέλετε να απαντήσω σε ερωτήσεις η μία από τις οποίες αφορά τις θεωρήσεις, το καθεστώς θεωρήσεων για Ευρωπαίους και Ρώσους πολίτες, ενώ το άλλο αφορά, η άλλη ερώτηση, αφορά τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας μετά την σύνοδο της Στοκχόλμης και την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ. Για αυτές τις δύο ερωτήσεις θέλετε να μιλήσω πρόεδρε, έτσι. Ωραία. Για το θέμα των θεωρήσεων, το Συμβούλιο θέλει να σας υπενθυμίσει ότι το 2003 υιοθετήθηκε ένας κανονισμός που περιλαμβάνει ένα ειδικό ε, ε, έγγραφο διέλευσης και ένα απλοποιημένο έγγραφο διέλευσης. Μετά από τρία έτη, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η θέση σε ισχύ του συστήματος αυτού προχωρούσε άνετα, χωρίς προβλήματα και ότι οι δύο πλευρές ήταν ικανοποιημένες. Σε ένα πιο μακροπρόθεσμο πλαίσιο προοπτικής, σας μιλώ για την περιοχή του Καλίνιγκραντ και την υπόλοιπη ρωσική ομοσπονδία. Το καθεστώς ε, απλοποιημένης διέλευσης όπως αποκαλείται εξαρτάται από την μελλοντική σύναψη συμφωνιών μεταξύ Ένωσης και Ρωσικής Ομοσπονδίας συνολικά. Σε μια κοινή δήλωση που εκδόθηκε μετά το Συμβούλιο Σύνδεσης Ένωσης Ρωσίας για θέματα Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων τη 2 Δεκεμβρίου, της Δεκεμβρίου του 2009, οι συμμετέχοντες αποφάσισαν να συζητήσουν πιθανές τροποποιήσει τη συμφωνία ε, με τη Ρωσία για τη διευκόλυνση των θεωρήσεων για να γίνει πιο εύκολη, εύκολες μετακινήσεις Ευρωπαίων πολιτών και Ρώσων πολιτών. Ιδιαίτερα δε ε, ε, μετακινήσεων κατοίκων της περιοχής του Καλίνιγκραντ. Με την ίδια κοινή δήλωση η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ρωσία ήθελαν να διαμορφώσουν ε, συμφωνίες διέλευσης με, με τις γειτονικές χώρες που μπορεί να ενδιαφέρονται. Στο πλαίσιο αυτό ο κανονισμός 1825 του 2006 του Συμβουλίου και, του, και της Επιτροπής για, και του Κοινοβουλίου για την ε, μορφή, για την ε, τροποποίηση των, των, ε, του κεκτημένου Σέγγεν και που επιτρέπει την συμβουναψή συμφωνιών με γειτονικέ τρίτε χώρε για την εφαρμογή του καθεστώτο ε, απλοποιημένη διασυνοριακή διέλευση υιοθετήθηκε χωρί πρόβλημα. Είναι ένα θέμα ωστόσο αυτό που ανοίγει στα κράτη-μέλη που αφορά ο εν και την Ρωσία. Το Συμβούλιο καταγράφει ότι συνεχίζονται διαπραγματεύσει μεταξύ Λιθουανία και Ρωσία και μεταξύ Πολωνία και Ρωσία για τον σκοπό αυτό. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση για τις στρατηγικές σχέσεις Ένωσης Ρωσίας το Συμβούλιο υπογραμμίζει ότι μετά τη σύνοδο κορυφή με τη Ρωσία που έλαβε χώρα στη Στοκχόλμη τον περασμένο Νοέμβριο κατά τη διάρκεια τη Ισπανική Προεδρία θα υπάρξει και άλλη μια σύνοδο κορυφή με τη Ρωσία, στη Ρωσία αυτή τη στιγμή, αυτή τη φορά. Θα δοθεί μια όθηση στι σχέσει και από τι δύο πλευρέ. Όπω είναι λογικό, πάντα μπορεί να υπάρχουν δυσκολίε που να σχετίζονται με το σύνθετο χαρακτήρα των σχέσεων, υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, αλλά η σχέση μεταξύ Ένωσης και Ρωσίας είναι πολυμερής, εκτεταμένη, συνδέεται με αυξανόμενα οικονομικά και εμπορικά, με αυξανόμενες εμπορικές και οικονομικές σχέσεις. Υπάρχει μια μεγάλη αλληλεξάρτητη στον τομέα της ενέργειας, υπάρχουν κοινά συμφέροντα σε άλλους τομείς, όπως τομείς που ξεπερνούν και τις χώρες μας μερικές φορές και προκλήσεις οικουμενικού μερικές φορές χαρακτήρα που θα έπρεπε να αντιμετωπίσουμε όσο πιο ε, ενιαία γίνεται. Πάντα λοιπόν θα είναι θετικό να αναζητούμε τρόπους για να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με τη Ρωσία διατηρώντας ωστόσο σταθερές τις θέσεις μας σε ό,τι αφορά τις αρχές και τις αξίες που προασπίζει η Ένωση. Σε ό,τι αφορά την προσχώρηση της Ρωσίας στον ΠΟΕ, η Ένωση υποστηρίζει μια τέτοια ένταξη, ωστόσο η Ρωσία είναι αυτή που να τα μέτρα για να ενταχθεί στον οργανισμό αυτό. Σε ό,τι αφορά τη νέα συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας, και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι θα ήταν καλό να υπάρξει μια νέα διευρυμένη συμφωνία. Η Συμφωνία Εταιρική Σχέση και Συνεργασία μεταξύ Ένωση και Ρωσία ε, που συνάφθηκε στη δεκαετία του 90 είναι πλέον παροχημένο σε πολλέ διαστάσεις του. Άλλαξαν πολλά πράγματα από τη δεκαετία του 90. Χρειάζεται να προχωρήσουμε προ μια νέα συμφωνία Είμαστε φιλόδοξοι. Έχουμε θέσει τον πύχη ψηλά. Θέλουμε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε όλου του τομεί συνεργασία Ένωση Ρωσία. Υπήρξε πρόοδο σε κάποιου τομεί στι διαπραγματεύσει. Άλλοι τομεί πάνε πιο αργά. Επενδύσει σε εμπόριο. Για μας πάντω είναι πολύ σημαντικό να υπάρξουν κάποιε στέρεε συμφωνίε με τη Ρωσία στον τομέα του εμπορίου, των επενδύσεων και τη ενέργεια. Σε ό,τι αφορά το καθεστώς ελεύθερων συναλλαγών, συμφωνούμε να υπάρξει μια συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών, ελεύθερου εμπορίου, όταν η Ρωσία γίνει, γιατί μόνο έτσι γίνει αυτό το γεγονό, μέλος του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπόριου. Σε ό,τι αφορά την απελευθέρωση των θεωρήσεων, πρόκειται για ένα θέμα που έχει πολύ μεγάλη πολιτική σημασία και επηρεάζει ευθέως τους πολίτες και τις ουσίες και της Ένωσης. Θα ήθελα να πω ότι συμμεριζόμαστε την πρόθεση να υπάρξει μια διευκόλυνση στις θεωρήσεις. Θα ήταν μάλιστα ιδεώδης να υπάρξει και μια κατάργηση των θεωρήσεων, αλλά μέχρι να γίνει αυτό έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, ενώ επιπλέον πρέπει να υπάρξει εξισορρόπηση των αξιών που διακυβεύονται ασφάλειας και να γίνεται πάντα βάση της αρχής της αμοιβαιότητας. Σε ό,τι αφορά την Ουκρανία, τη Μολδαβία και τη Γεωργία, κάθε μία από τις χώρες αυτές είναι διαφορετική, έχουν ε, διαφορετική ένταση σε ό,τι αφορά τις θεωρήσεις δεν μπορούμε να πούμε λοιπόν πώς θα πρέπει αυτή τη στιγμή να προχωρήσουν, να ενταχθούν οι χώρες αυτές εδώ στο διάλογο για τις θεωρήσεις που έχουμε με την Ρωσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Θα πάρω τώρα τις δύο συμπληρωματικές ερωτήσεις από τον κύριο Πάντα και τον κύριο Πόσελτ. Του κύριο Πάντα πρώτος. Ο, κύριος Πόσελτ. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση για τα δύο πολύ κρίσιμα θέματα όσον αφορά τη δημοκρατία, το κράτο δικαίου, τα ανθρώπινα δικαιώματα. Εκεί παρουσιάζονται τα μεγαλύτερα ελλείμματα και πόσο ελληματικό είναι ο διάλογο σε αυτά τα τόσο κρίσιμα θέματα. Γιατί έχουμε εδώ την αίσθηση ότι οι εξελίξει πάνε προ τα πίσω και όχι προ τα μπρο. Αυτό ήταν το ένα. Το δεύτερο, ενεργειακή ασφάλεια. Τι ακριβώ γίνεται με τι ε, ενεργειακέ διαπραγματεύσει. Κύριε Υπουργέ. Κύριε Βουλευτά, μία από τις προτεραιότητες και τους στρατηγικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ασφάλεια εφοδιασμού, ε, η ενεργειακή ασφάλεια, κυρίως όσον αφορά τον εφοδιασμό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και κυρίως ε, μετά την κρίση του αερίου, αυτή η κρίση που υπήρξε στις αρχές του 2009 ανάμεσα στην Ουκρανία και τη Ρωσία, όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατανόησαν τη μεγάλη σημασία του, της ασφάλειας ε, του ενεργειακού εφοδιασμού. Ο στόχος λοιπόν της ενεργειακής ασφάλειας είναι ένας από τους ε, βασικότερους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει βέβαια και άλλο ένα σημαντικό στόχο που είναι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Όσον αφορά λοιπόν στην, ε, στον ε, ενεργειακό εφοδιασμό, το ε, Συμβούλιο τονίζει ότι είναι απαραίτητο να έχουμε μια μεγαλύτερη διαφοροποίηση των πηγών αλλά και μεγαλύτερη διαφοροποίηση των προμηθευτών και των διόδων παροχής. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει να ανοίξει περισσότερο η βεντάλια των δυνατοτήτων, να προσπαθήσουμε να αποφύγουμε μορφές ολιγοπολείο ή υπερβολικής εξάρτησης. Αυτό που σημαίνει σε πολλά κράτη-μέλη που έχουν την ενεργειακή εξάρτηση από τη Ρωσία, αλλά είναι σημαντικό η εξάρτηση αυτή να μην καταστεί υπερβολική. Και ας μην ξεχνάμε ότι η Ευρώπη για μεγάλο χρονικό διάστημα του προηγούμενου αιώνα ήταν διαιρεμένη. Έτσι, αυτό λοιπόν σημαίνει ότι κάποιες σχέσεις ε, ε, στον ενεργειακό τομέα εξακολουθούν ακόμα να υφίστανται. Η κρίση λοιπόν των ε, αρχών του αιώνα αυτού κατέστησε σαφές ότι ορισμένες χώρες που δεν επλήγησαν από την κρίση μπόρεσαν να δείξουν αλληλεγγύη απέναντι σε άλλες χώρες γιατί όπως σας είπα υπήρχε αυτή η σχέση μεταξύ τους. Κατόπιν τούτου καταλαβαίνετε ότι οι σχέσεις είναι πολύ σημαντικές. Εμείς είμαστε αναμφισβήτητα υπέρ της διαφοροποίησης των ενεργειακών πηγών και είμαστε επίσης υπέρ του ότι ε, αγωγοί όπως ο Ναμπούκο, προγράμματα όπως το South Stream να προχωρήσουν έτσι ώστε να προκύψουν ε, δυνατότητες που αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν. Όσον αφορά λοιπόν αυτούς ε, τους στόχους, οι στόχοι αυτοί πρέπει να διευκολυνθούν και διευκολύνονται μέσα από τις συνθήκες Λισαβόνα, γιατί υπάρχουν στόχοι που κατά παρελθόν δεν υπήρχαν. Έτσι λοιπόν μέσω των στόχων αυτών είναι απολύτως απαραίτητο να υπάρχει στρατηγική συνεργασία με τη Ρωσία ακόμα και σε ε, ενεργειακό επίπεδο, προφανώς και σε άλλα επίπεδα η συνθήκη της Λισαβόνας μεταξύ άλλων ενισχύει την εξωτερική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει πλέον ο ή, αρμοστής της Ευρωπαϊκής Ένωσης η ύπατη αρμοστής, άρα δηλαδή η ε, συνθήκη της ε, Λισαβόνας ε, πλέον διευκολύνει τη ζωή μας σε πάρα πολλούς τομείς στις διαπραγματεύσεις και για το ενεργικό θέμα και με τη Ρωσία και με άλλους εταίρους. Αυτό λοιπόν είναι το σκηνικό που μπορώ να σας παρουσιάσω όσον αφορά τη σχέση με τη Ρωσία. Δηλαδή διαπραγματευόμεθα επί ενός συμφώνου όπου το ενεργειακό είναι καθοριστική σημασία. Οι διαπραγματεύσεις για αυτήν την συμφωνία έχουν προχωρήσει. Οι προοπτικές είναι πάρα πολύ καλές, αλλά προφανώς είναι μια συμφωνία που είναι περίπλοκη, που ακόμα θα ακολουθήσουν αρκετές διαπραγματεύσεις. Πέρα από όλα αυτά ε, υπάρχει και μία πρόοδο που πρέπει και αυτή να εξυγχρονιστεί, να επικαιροποιηθεί. για τελευταία χρόνια έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Η Ρωσία είναι προφανώ μία από τι χώρε που έχουν αλλάξει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και αυτό είναι κάτι που πρέπει να έχουμε κατά νου. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Έχω ερωτήσεις από άτομα που δεν έλαβαν μέρος στη συζήτηση και αυτές θα είναι και οι δύο τελευταίες, διότι νομίζω ξεπεράσαμε κατά πολύ την ώρα. Σόνικ και ο κύριος Σόνικ και η κυρία Ζέμκο. Ο κύριος Σόνικ πρώτος. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σχετικά με την ερώτηση 9 που επρόκειτο να υποβάλω εξ ονόματος της κυρίας Αντρικένε θα θέλω να αναφερθώ στον ε, πυρηνικό σταθμό που πρόκειται να κατασκευαστεί κοντά στα σύνορα. Μετά από την εμπειρία του Τσερνομπίλ γνωρίζουμε πόσο παρακινδυνευμένο είναι αυτό. Πρόκειται το Συμβούλιο να θέσει το θέμα στις συνομιλίες. Ευχαριστώ επειδή αυτή η ερώτηση αναφέρεται στην προηγούμενη, στο προηγούμενο θέμα, θα αφήσω τον Υπουργό να κρίνει. Τώρα, περνάμε στις ερωτήσεις 7 και 8. Θα ήθελα να επανέλθω στην... Ε, επανέρχομαι σε ερωτήσεις 7-8 που αφορούν τις σχέσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Ο Υπουργός πολύ σωστά είπε ότι οι σχέσεις πρέπει να στηρίζονται σε κάποιες αξίες. Αν ισχύει αυτό, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει δικέ υποχρεώσει για έναντι εκείνων που αγωνίζονται για τα ανθρώπινα δικαιώματα στη Ρωσία. Η ερώτησή μου είναι εξή. Στην πολιτική των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση, υπέρ των υπέρμαχων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Ρωσία δεν θα έπρεπε να βοηθήσουμε αυτά τα άτομα στο πλαίσιο τη σχετική πολιτική, ώστε να μπορούν αυτοί οι υπέρμαχοι των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να αποκτήσουν θεώρηση βίζα πιο εύκολα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ. Minister, if you are ready. Είστε έτοιμος, σας δίνω το λόγο. Σε ό,τι αφορά την ερώτηση για την πυρηνική ασφάλεια, πρέπει να σας πω ότι η ευθύνη για την πυρηνική ασφάλεια που είναι εθνική εμπεριέχεται στις διεθνείς συμφωνίες του Διεθνούς Οργανισμού Πυρηνικής Ασφάλειας, του ΟΗΑ, όπου είναι συμβαλόμενα μέλη η Λευκορωσία, η Ρωσία, η ευρωτόμη και τα περισσότερα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το Συμβούλιο θεωρεί ότι τα συμβαλόμενα μέρη που είναι κοντά σε έναν πυρηνικό σταθμό πρέπει να μπορούν να μετέχουν, στις, να ενημερώνονται πλήρως γιατί μπορεί να επηρεαστούν. Η συμφωνία λοιπόν Ευρατόμ Ρωσίας που ασχολείται με τις ε, ειρηνικές εφαρμογές της πυρηνικής ενέργειας μπορεί να περιλάβει, ε, περιλαμβάνει διατάξεις για τις ε, απαιτήσει ελέγχου πυρηνικής ασφάλειας. Να σας υπενθυμίσω επίση ότι το θέμα αυτό αντιμετωπίζεται σε περιοδική βάση στα πλαίσια του διαλόγου Ένωσης Ρωσίας στον τομέα της ενέργειας. Σε ό,τι αφορά την αξιολόγηση των συνεπειών σε διεθνέ πλαίσιο, το Συμβούλιο παρατηρεί ότι η Λευκορωσία είναι τμήμα της συμφωνίας του ΕΣΠΟ για την αξιολόγηση του αντίκτυπου στο περιβάλλον των πυρηνικών σταθμών που έχει δεσμευτικές ε, προϋποθέσεις για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και των, ε, ε, επιπτώσεων ευρύτερα στο περιβάλλον. Ωστόσο, εν πολλής, ε, το, η συμφωνία του ΕΣΠΟ λέει ότι οι υπεύθυνοι για την περιβαλλοντική μελέτη είναι οι κατασκευαστές του σταθμού. Η Ρωσία δεν είναι μέλος της συμφωνίας αυτής. Εμείς θα θέλαμε να εφαρμόσει η Ρωσία σε θελούσια βάση τη συμφωνία του ΕΣΠΟ. Κάτι που κάνει εδώ και καιρό σε ό,τι αφορά τους πυρηνικούς σταθμούς που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Εν τέλει, σε ό,τι αφορά την ερώτηση του κυρίου βουλευτή για το θέμα των δικαιωμάτων του ανθρώπου και τη Ρωσία. Είχαμε μια προηγούμενη συζήτηση για θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων εδώ στην Ολομέλεια και πιστεύω ότι τα κριτήρια για την υποστήριξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την καταγγελία των παραβιάσεών τους ισχύουν για οποιαδήποτε περιοχή του κόσμου ανακύψουν. Ε, με κάθε δικαίωμα και με υποχρέωση θα έλεγα η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και πρέπει να καταγγείλει παραβιάσεις που και εμείς κάνουμε θα πρέπει να κάνουμε όταν υπάρχουν τέτοιε παραβιάσεις στο ιστορικό τη Ένωση. Η σύνδεση τέτοιων καταγγελιών με την πολιτική θεωρήσεων είναι ένα άλμα που αυτή τη στιγμή πολύ δύσκολο μπορούμε να συγκεκριμενοποιήσουμε. Γίνεται μία αυτή τη στιγμή ευρεία εκτεταμένη συζήτηση για θέματα θεωρήσεων Δεν νομίζω ότι στο πλαίσιο αυτό μπορεί να υιοθετήσει κάποιο συγκεκριμένους δρόμους για την διευκόλυνση των θεωρήσεων. Όπως λέω ωστόσο, έχουμε μια γενική συζήτηση για το θέμα των διαπραγματεύσεων θεωρήσεων με τη Ρωσία και εκεί νομίζω πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας. Τις θεωρήσεις εν γέννη, διότι εκεί μπορεί να έχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα σε ό,τι αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία των ατόμων και την βελτίωση, την αύξηση των δυνατήτων, ούτως ώστε η Ευρώπη να περάσει τις αξίες της και να επιτρέψει και σε πολίτες άλλων χωρών εκτός Ένωσης να ε, εκμεταλλευτούν τις δυνατότητες αυτές. Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σα, κύριε Υπουργέ. Οι ερωτήσει που δεν απαντήθηκαν λόγω έλλειψης χρόνου θα απαντηθούν εγγράφως. Λύεται η συνεδρίαση. Απλώς <clears throat> θέλω να κάνω μια ανακοίνωση. Η, η, ομάδα του ΕΛΚ, οι χριστιανοδημοκράτε, οι σοσιαλιστέ μου έχουν υποβάλει αιτήσει για διορισμούς στις αντιπροσωπείες και τις επιτροπές εάν δεν λάβουμε σχόλια πριν την, απόφαση, πριν την έγκριση των πρακτικών αυτοί οι διορισμοί θα γίνουν δεκτοί η επόμενη συνεδρίαση θα